Λέξουν και άλλες πολιτικές ομάδες. Η πρόεδρος λέει δεν χρειάζεται να μου κάνετε έκκληση διότι έτσι θα προχωρήσουμε. Προχωρούμε λοιπόν στις ψηφοφορίες, έληξη συζήτηση. Για την Κένια λοιπόν και την αποτυχημένη σύλληψη του Σουδανού Προέδρου Ομάρ Ελμπεσίρ. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έξι προτάσεις ψηφίσματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία και ειδικότερα στην περίπτωση του Χαϊτάν Αλμαλέχ. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Έχω κάποιες ανακοινώσεις να κάνω. Εν τω μεταξύ όμως να δώσω το λόγο στην κυρία Γκέπχαρτ. Με συγχωρείτε, δεν ε, έβαλα γέρο στην κάρτα μου, αλλά έχω υπερψηφίσει το ψήφισμα. Το σημειώνουμε, ευχαριστώ. Έχω λάβει λοιπόν την θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Κυρία Έρκ, παρακαλώ. Δεν δούλεψε το μηχάνημά σας για την ψηφοφορία. Το σημειώνω. Άλλος. Προχωρώ λοιπόν στα